Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να μην είμαστε ακόμα σε απαρτία, αλλά παρευρίσκονται οι συντονιστές, οπότε και μπορούμε να αρχίσουμε. Θα προεδρεύσω σύντομα μέχρι να έρθει ένας αντιπρόεδρος κάποια στιγμή. Και πάμε στην ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη όπως έχει κατατεθεί. Ε, μία μικρή παρατήρηση, το σημείο 12 να βάλετε για την επόμενη φορά, εάν δεν έχετε αντιρρήσεις. Ωραία. Άλλη ανακοίνωση. Όπως πάντα, η παρούσα συνεδρίαση μεταδίδεται απευθείας στο διαδίκτυο. Επίζω να έχετε και να έχουμε πολλούς ακροατές όσο και θεατές. Ε, Μετά στις 26 και 27 Αυγούστου μετέβει η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Ελλάδα. Έχετε την έκθεση στα αγγλικά. Αλλά βεβαίως η έκθεση αυτή υπάρχει και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Επίσης έχετε στα χέρια σας τα πρακτικά της 5 η Σεπτεμβρίου. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης θα θεωρούνται θα θεωρηθούν μάλλον εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ερχόμαστε λοιπόν στον προσκεκλημένο μας και χαιρόμαστε που βλέπουμε τον Επίτροπο κύριο Νέβεν Μίμητσα. Καλώς ορίσατε. Έχετε μέσα στο λόγο. Παρακαλώ. It's a really valuable occasion today. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή και πολύ χρήσιμο πιστεύω που θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε πού βρισκόμαστε τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου. Την ανάληψη του χαρτοφυλακίου για, τις, ε, για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο για να ε, υλοποιήσουμε την ατζέντα για τον καταναλωτή, αν και περιμέ... αναμένουμε και κάποια σημαντικά βήματα τους επόμενους μήνες. Θα είναι η κύρια μου προτεραιότητα στις επόμενους ε, μήνες. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ολοκληρωθούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, τα φάκελοι που αφορούν στην ασφάλεια των προϊόντων, τα ιατρικά εργαλεία και τις, ε, τους λογαριασμούς πληρωμής. Εγώ θα ήθελα και οι τρεις αυτοί φάκελοι να ολοκληρωθούν στην ε, τρέχουσα νομοθετική περίοδο. Ο νέος κανονισμός για την ασφάλεια των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς έχει μεγάλη σημασία για να βελτιωθεί το γενικό πλαίσιο και η ε, παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων. Είμαι ε, ευτυχής και θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την Προεδρία του Συμβουλίου, που έδωσαν ε, την απαιτούμενη έμφαση και προτεραιότητα στο θέμα αυτό και έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε σημαντικά τι ε, διαπραγματεύσεις και τον τριμερή διάλογο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τον κύριο Σάντελ Μόζε και την κυρία Πιέτη Κάινεν. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση στο ζήτημα της ε, χώρας προέλευσης. Θα Επίσης ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε την δημιουργία του συστήματος RAPEX, της άμεσης και γρήγορης ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα. Είναι σημαντικό αυτό το σύστημα για να ανταλλάσσονται τέτοιες πληροφορίες. Και τώρα έρχομαι στις δύο ε, προτάσεις ε, νομοθετικές ε, για τους, τα, τα, τα ιατρικά υλικά. Ο πρωταρχικός μας στόχος εδώ είναι να διασφαλίσουμε την ε, δημόσια υγεία και την ασφάλεια ε, των ασθενών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εσωτερική αγορά και την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ιατρικών Εργαλείων και Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το, για το έργο σας και ιδιαίτερα τον εισηγητή, την κυρία Μπέρα προχωρήσουμε ε, με αποφασιστικότητα στην οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμής. Ακόμα και σήμερα 58 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, άνω των 15 ετών δεν έχουν πρόσβαση σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Πολλές φορές οι πολίτες αναγκάζονται να πληρώνουν πέρον κατέλη τραπεζικά ή αναγκάζονται να αποκρυπτογραφούν πολύ δύσκολους τραπεζικούς όρους η Επιτροπή ΙΜΚΟ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στον τομέα αυτό, σε αυτήν την πρόταση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέπχαρτ για την, το προσχέδιο έκθεσης ε, και τη συνεργασία που είχαμε και η οποία μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε το έργο μας σε αυτόν τον τομέα ε, γρήγορα. Η δεύτερη προτεραιότητά μου είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση των ήδη ε, υιοθετημένων εγκεκριμένων νόμων νομοθεσίας. Θα είμαι αποφασισμένος να εργαστώ προκειμένου η νομοθεσία που αφορά στην εναλλακτική ή online επίλυση συγκρούσεων και διαφορών να υλοποιηθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορο γίνεται. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο το οποίο να λειτουργεί σωστά και να είναι φιλικό προς τον χρήστη μέχρι το τέλος του 2016. Προσπαθώ επίσης να αναλάβω με δική μου πρωτοβουλία ε, βήματα για το ζήτημα της ε, συλλογικής αποζημίωσης. Ακόμα και αν η νομοθετική πρωτοβουλία εδώ, η συλλογική αγωγή, συλλογική προσφυγή δεν είναι ένα νομικά δεσμευτικό εργαλείο, θα ήθελα να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Και προς αυτήν την κατεύθυνση η Λουθανική Προεδρία στο Βίλνιους θα οργανώσει μια, ένα συνέδριο. Φασισμένος να ενισχυθεί η υφιστάμενη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή. Ιδίως όσον αφορά την εξάλληψη των αθέμητων εμπορικών ε, πρακτικών και την πλήρη τον πλήρη σεβασμό των ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή. Ήδη έχουν στη διάθεσή μας διάφορα σημαντικά εργαλεία και αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό, ένα από αυτά είναι για παράδειγμα το SWIB, ο, ο έλεγχος ε, των ε, ιστοσελίδων που γίνεται σε αιτήσια βάση, ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, και η συνεργασία και ο άμεσος διάλογος με τη βιομηχανία έτσι ώστε να ε, υπάρξουν άμεσες βελτιώσεις σε διάφορους τομείς μέσω της εθελοντικής συνεργασίας. Όμως πρέπει να βελτιώσουμε κάποια ε, σημεία έτσι ώστε η δράση με την προστασία του καταναλωτή να είναι ε, ακόμα πιο αποτελεσματική και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές οι καταναλωτές ε, βασίζονται στις γνώμες που εκφράζουν ε, άλλοι καταναλωτές, για παράδειγμα στον τομέα των ξενοδοχείων. Γνωρίζουμε όμως ότι πολλές φορές αυτές οι, αυτές οι απόψεις άλλων καταναλωτών στην πραγματικότητα είναι ψεύτικες. Και αυτό, αυτές εκτιμώνται μέχρι και το 30% να ε, είναι μη αληθινές. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο σε αυτόν τον τομέα. Και έχω ξεκινήσει να προετοιμάζω μια έκθεση και την οποία ε, του χρόνου θα παρουσιάσω στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε σχέση με έναν κανονισμό για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Προετοιμάζοντας αυτή την έκθεση θα ξεκινήσουμε σύντομα μία δημόσια διαβούλευση. Είναι μια διαδικασία στην οποία θα ήθελα να και ευελπιστώ ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν ε, χωρίς περιορισμούς και θα μπορέσουν να μας δώσουν ιδέες για το ποιες είναι οι βέλτιστες λύσεις για να δημιουργήσουμε ένα μακροπρόθεσμο ε, πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή στην Ευρώπη και των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Θα ε, ήθελα να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαρίστω να έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων επί του ζητήματο αυτού με την Επιτροπή σα. αν το επιθυμείτε. Κυρία Πρόεδρε, τα μέλη. Σημαντικότερη προτεραιότητά μου είναι να έχουμε απτά αποτελέσματα στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Επίτροπο Έντιγκερ και θα παρουσιάσουμε από κοινού στον επόμενο φόρουμ ε, πολιτών για την ενέργεια μία έκθεση για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και πώς ε, μπορούν να βοηθηθούν οι καταναλωτές για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειάς τους. Συνεργαζόμαστε επίσης και με τα κράτη-μέλη στο ζήτημα της ε, ενέργειας. Είχαμε ήδη πολύ ενθαρρυντικές πρωτοβουλίες και θα ήθελα να δω εάν αυτές μπορούν να εξαχθούν και να αναλυθούν και από άλλα κράτη-μέλη όλα αυτές οι πρωτοβουλίες που σας ανέλησα βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, σε στοιχεία. Έχουμε ζητήσει μελέτες στον τομέα, για παράδειγμα, της ηλεκτρικής ενέργειας, στη ε, συμπεριφορά των καταναλωτών, για θέμητες ή παραπλανητικές ε, τακτικές, για την προστασία των παιδιών καταναλωτών. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, πράγματι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και ευελπιστώ ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί αμύωτη και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτροπε, για τις εξηγήσεις και τις περιγραφές. Ουσιαστικά μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι αυτό το πρόγραμμα, μέχρι τις ευρωεκλογέ. Θα ήθελα να ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Πρώτα οι συντονιστές με τους κυρίους Φαπ πρώτα και μετά ε, Την κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να σα πω καταρχά ότι χαιρόμαστε που βρήκατε χρόνο μετά το καλοκαίρι να έρθετε να μα ενημερώσετε για τις σκέψεις σας ως προς ε, τη μετεξέλιξη και ολοκλήρωση της εσωτερική αγορά, ω προς το θέμα των καταναλωτικών αγαθών και την προστασία των καταναλωτών. Ειλικρινά, θα με ενδιέφερε λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας Πώς βλέπετε τα πράγματα και πώς συνεργάζεστε με τους όλους τους συναδέλφους και τις άλλες γενικές διευθύνσεις και πώς έχετε συντονιστεί ως καταποκλειστικότητα αρμόδιος για την προστασία καταναλωτών. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων που είναι στη δική μας επιτροπή. Μιλήστε και για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά εμείς πηγαίνουμε και για ε, θέματα σήμανσης, τα γενικά καταναλωτικά αγαθά. Ε, και σας ερωτώ τα εξής δύο. Πρώτον, το Κοινοβούλιο στη ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα του ελέγχου και της προστασίας ε, του ε, ασθενούς. ισορροπία ανάμεσα στα ασφαλιστικά ταμεία από τη μια ε, και στην καινοτομία της βιομηχανίας από την άλλη. Γιατί ε, όταν μια φορά έχουν κακέ εμπειρίε. Μπορεί να αφορά αυτό ένα καταναλωτή με μονομένου, αλλά οι περισσότεροι ασθενεί και καταναλωτέ εποφελούνται πάρα πολύ από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και χαίρουν μεγάλη εκτίμηση στα μάτια του αυτά. Και μετά, κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στην υλοποίηση στα κράτη-μέλη, στην εφαρμογή, του λεγόμενο enforcement. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και τις επόμενες μέρες θα τα βρούμε μπροστά μας όταν θα ψηφίσουμε την, ε, ασφάλεια, την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων γενικά. Έχει να κάνει αυτό με το σήμα ε, προέλευσης, το Made In. Ε, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη, χωρίς μελέτη σκοπιμότητας, έχει εισαγάγει κάποιες διατάξεις στην οδηγία αυτή Εσεί θα ήσασταν πρόθυμο να συζητήσετε με τον κύριο Πούλιο μεγαλύτερη και ευρύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Και τη μικρομεσαία, αν μου επιτρέπετε, κυρία Βάιλερ, γιατί στη Γερμανία γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Η κυρία Γκέμπχαρτ, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μίμητσα για την ενημέρωση. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό το γεγονός ότι εδώ και λίγο καιρό έχουμε τροπό που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα προστασίας των καταναλωτών. Και αυτό κάνει καλό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ευεργετική επίδραση γιατί φαίνεται ότι έχει αναβαθμιστεί το θέμα. Και αυτό για μένα είναι πολύ καλό δήλωσα προθυμία να εργαστώ πάρα πολύ γρήγορα σε ό,τι αφορά τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί θα πρέπει το συντομότερο να φροντίσουμε στην παρούσα νομοθετική ε, περίοδο να ληφθεί κάποια απόφαση, διότι είναι πολλοί εκείνοι οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό γιατί δεν τους επιτρέπουν. Όχι ότι δεν θέλουν να ανοίξουν λογαριασμό, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, δεν θα τους αναγκάσουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να ανοίξουν ένα βασικό λογαριασμό για τις πληρωμές τους και δεν τους αφήνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σήμερα σχεδόν δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα ζει κάποιος χωρίς να έχει τραπεζικό λογαριασμό με τα διάφορα εμβάσματα που μπορεί να κάνει και πληρωμές ε, τραπεζικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε αυτός ο βασικός λογαριασμός πληρωμών να είναι δωρεάν ή αν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στοιχειώδη συμβολικά τραπεζικά τέλη ε, να χρεώνονται. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχω απογοητευτεί λίγο από αυτά που μας είπατε για τις συλλογικές ε, αγωγές. Εμείς ως Κοινοβούλιο το συζητούμε αυτό εδώ και χρόνια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ και χρόνια μας Ταζουν διάφορες μελέτες, τις οποίες κάνουν κιόλα, αλλά ελέγχουν τη μελέτη, ξαναελέγχουν την άλλη μελέτη και τώρα λέτε πάλι θα το ε, ε, επανελέγξετε. Ναι, να βαθούμε και στο διατάφτα. Είτε θα μας πείτε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το θέλουμε, που είναι και αυτό καθαρή εξήγηση και θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε στο Κοινοβούλιο, ε, είτε θα μας πείτε το θέλουμε, αλλά φέρτε μια πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να το αναβάλουμε στο διηνικές. Ναι, να το μελετήσουμε, να το ελέξουμε, θα κάνουμε κάτι, το προετοιμάζουμε, αυτό δεν μας ικανοποιεί. Και σας παρακαλώ, ειλικρινά, να πιέσετε λίγο περισσότερο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν συμφωνούν όλοι, ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν οι πάντες για αυτό το θέμα. Παρά όλα αυτά οι πολίτες χρειάζονται απάντηση για το τι μέλη γενέστε. Και δεν μπορούμε να του αφήνουμε σε αυτή την αβεβαιότητα. Και ένα τρίτο και τελευταίο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η χώρα προέλευσης ε, για τα προϊόντα, έτσι, το made in, πού παράγεται ένα προϊόν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και εδώ χρειαζόμαστε μια λογική απάντηση. Πολλοί είναι εκείνοι οι πολίτες που θα ήθελαν να γνωρίζουν το προϊόν που αγοράζουν ή που επιθυμούν να αγοράσουν, που έχει κατασκευαστεί, με ποιες προϋποθέσεις και ποιους όρους. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που διαφορούν, αλλά υπάρχουν επίσης πολλοί που ενδιαφέρονται. Και εδώ χρειάζεται κάποια ένδειξη. Μια ένδειξη που να έχει και νόημα και να θέλει να πει και κάτι το λέω υπερβολικά γιατί δεν ισχύει αυτό απλώς, αλλά το λέω έτσι υπερβολή. να ράβετε κάπου ένα ποκάμισο και να έρχεται στη Γερμανία, του βάζουν τα κουμπιά και να γράφει Made in Germany. Ενώ έχουν ραφτεί μόνο ε, τα ε, κουμπιά στη Γερμανία και ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Το ξέρω ότι δεν θέλουν να επιβαρύνονται ιδιαίτερα, ούτε εμεί θέλουμε να του επιβαρύνουμε, αλλά να γνωρίζουν οι πολίτε περί τίνο πρόκειται για να μπορούν να ψωνίζουν και με τα λόγου γνώσεω, στο βαθμό που το επιθυμούν, λέω. Ευχαριστώ. vielen Dank. Ähm, ich äh, den Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω την Προεδρία στον κύριο Κοφεράτη, να κάνω δύο σύντομες ερωτήσεις ή σχόλια. Πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ε, πραγματικά μεγάλη κατανόηση για το γεγονός ότι θέλουμε να ολοκληρωθούν οι τρεις εκκρεμούσες οδηγίες πριν τις εκλογές για να ε, αρχίζουν να ελοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σωστό αυτό και απολύτως θεμητό. Και του χρόνου θα δοθεί ιδιαίτερη ε, έμφαση, λέτε, στην εφαρμογή. Γιατί πραγματικά αυτό χωλαίνει παντού, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Και θέλω να πω τα εξής που με ανησυχούν και μένα λίγο. Το πρώτο είναι συλλογικές αγωγές. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω πώς μπορείτε να το εξηγήσετε περισσότερο, από όσα άκουσα να μας λέτε, ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σας υποστηρίζουν αρκετά να πάτε μέσω των κρατών μελών, γιατί κάνετε διάσκεψη στη Λιθουανία, δεν ξέρω και μετά. Προσπαθείτε δηλαδή μέσω των κρατών μελών να ε, τα κερδίσετε τα κράτη στην προσπάθεια αυτή στο πλευρό σας. Το κατανοώ και ευφυής δρόμος είναι αυτός, αλλά έχουμε και εμείς την εμπειρία που λέει ότι τα κράτη-μέλη μπλοκάρουν ακόμα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και από κάποιους συναδέλφους από ε, άλλες ομάδες. Και ε, όλο και κάποια χώρα θα έχει εκλογές πάντα. Νομίζω θα πρέπει να εμπιστευτείτε και τους συμμάχους σας, αν μη τι άλλο, ε, ε, αυτή είναι ένα μεγάλο τμήμα του Κοινοβουλίου και η δική μου πολιτική ομάδα αλλά και άλλοι και θυμάμαι κάτι που είχα διαβάσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται και ένα τρίτο δρόμο, δηλαδή όχι το αμερικανικό σύστημα αλλά ούτε και το status quo που επικρατεί αυτή τη στιγμή, αλλά επεξεργάζονται ε, στην ουσία της μια νέα πρόταση. Και ένα τελευταίο, ε, πολύ καλό, ε, η διαφάνεια στη δημολόγηση της ενέργειας, όχι μόνο στη δική μου χώρα, παντού στην Ευρώπη. Νομίζω τα τιμολόγια της ενέργειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα στο μέλλον. Και αυτό είναι το α και το ω για να αλλάξει οτιδήποτε ή διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα τιμολόγια. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και εθνικές και ευρωπαϊκές και καλό θα ήταν να φέρετε εκεί κάποια διαφάνεια και θα σας υποστηρίξουμε. Και αν μπορείτε να το κάνετε αυτό πριν τις ευρωεκλογέ θα ήταν ευχή έργων. Διότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να αποδείξουν ε, πολλοί συνάδελφοι ότι ορίστε η Ευρώπη σε αυτό το θέμα που μας θίγει στην καθημερινότητά μας και στο πετσί μας όλους τους πολίτες δραστηριοποιείται. Σας ευχαριστώ πολύ και να έρθει ο κύριος Κοφεράτη να προεδρεύσει. Θα σας ακούσω την απάντηση από τη θέση μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και πάλι εκφράσατε το μεγάλο σας ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Ε, αυτό το καταδεικνύεται εξάλλου από τις, στις δράσεις ε, της Επιτροπής σας. Ως προς την πολιτική προστασία ε, των καταναλωτών, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς έχει ε, ε, την καταπληκτική ευκαιρία να προωθήσει αυτές τις πολιτικές και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους. Κατά τη διάρκεια της ακρόας πρωτού κάνα να λάβω τα καθήκοντά μου εδώ στην Επιτροπή, προσπάθησα να τονίσω ότι είναι οριζόντια, εγκάρση αυτή η πολιτική προστασία των καταναλωτών. Τουλάχιστον 10 12 επίτροποι και οι άριθμες πολιτικές εμπλέκονται ε, στα θέματα των καταναλωτών. Αυτό που προσπαθούμε είναι σε πρόωρο στάδιο όταν εκπονούμε και συντάσσουμε σχέδια μελλοντικών νομοθετημάτων σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεκτιμούμε αυτή τη διάσταση ούτως ώστε οι καταναλωτές οι ίδιοι να καθοδηγούν ε, τρόπον την τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδηλώντας τις επιθυμίες τους. Μετά από δύο-τρεις μήνες που πέρασαν από την αρχή της θητείας μου, Uh, Από τη συνεργασία που είχα με άλλους επιτρόπους, επιβεβαιώθηκε αυτή η άποψή μου ότι ε, σε όλες τις πολιτικές ε, έχει σημασία η πολιτική των καταναλωτών. Παραδείγματος χάρη με την Αντιπρόεδρο Κρούς, Ε, ε, προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε από κοινού το, το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και ευελπιστώ ότι αυτό το πακέτο θα προσφέρει αυτά ωφέλη στους καταναλωτές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου. Το ίδιο ισχύει για τον Επίτροπο Μπαρνιέ Ε, για την οδηγία για το βασικό τραπεζικό λογαριασμό ή για τις τραπεζικές υπηρεσίες γενικότερα ε, για τις επιχειρήσεις, ε, για τη βιομηχανική πολιτική αντιπρόεδρος Ταγιάννη και ούτω καθεξής. Ένα από τα βασικά επιτεύγματα καλύτερα να μην κατηγορηθώ για υπερβολική εμπιστοσύνη, γιατί δεν είναι ένα επίτευγμα υπό την έννοια ότι έχει ήδη αλλά τουλάχιστον έχουμε ανοίξει το δρόμο πλέον για το ευρωπαϊκό εξάμεινο ούτω ώστε να εκφύγει του μακροοικονομικού δημοσιονομικού του πλαισίου και να ακολουθηθούν πιο ε, ειδικέ συστάσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντα των καταναλωτών, την κοινωνική πτυχή της οικονομικής ε, πολιτικής, της πολιτικής ανάκαμψης. Υπάρχουν τρία νομοθετικά πακέτα που επεξεργάζεται το Κοινοβούλιο και έχουν καταλητική σημασία. Είναι, ε, βρισκόμαστε σημείο καμπής για την έγκρισή τους από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Για τις ιατρικές συσκευές και τα ιατρικά, ε, ιατροφαρμακευτικά σκευάσματα, μάλλον για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, βλέπουμε αποφασιστικότητα και σπουδή από πλευράς του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ε, έχει την εντολή για τον τριμερή διάλογο Και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη ρότα τα κράτη-μέλη, ώστε το Δεκέμβρη, το αργότερα τον Ιανουάριο, να αρχίσει ο τριμερής διάλογος για το πακέτο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την ε, γενική ασφάλεια των προϊόντων. Έχω πλήρη επίγνωση ότι ζητήματα όπως η χώρα προέλευσης ή το σήμα προέλευσης ε, είναι το πρόσκομα για την έγκριση του πακέτου. Από πλευράς Επιτροπής θα ήθελα να τονίσω ότι πέρα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό του, της χώρας προέλευσης ε, στον ε, κοινό τελωνιακό κώδικα και το σχετικό κανονισμό, ε, και δυνάμει των κριτηρίων της τελευταίας ουσιαστικής μεταρρύθμισης του κοινού τελωνιακού κώδικα Ε, και ε, έχοντας ε, λάβει γνώση της θέσης του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών προκύπτει ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ή θα έλεγα αποκλίνοντας στρατόπεδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παίξει κέριο ρόλο στην προσπάθεια Ε, διεκπαιρέωση του Δήμους και έγκριση του σχετικού κανονισμού. Made in. Ε, για το σήμα προέλευσης, θεωρούμε ότι είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο που εντάσσεται στο πακέτο ασφάλειας για την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων και την ε, καταπολέμηση των επικινδύνων προϊόντων που ε, διατίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συλλογικές αγωγές και αποζημιώσεις είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε, που ανέφερα μάλλον και εγώ στην παρέμβασή μου, αλλά ανέφεραν επανειλημμένα και οι συντονιστές. Εκρεμεί εδώ και πολύ χαιρό το ζήτημα. Ε, οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, ζητούν ένα πιο ισχυρό νομοπαρασκευαστικό ρόλο, δηλαδή ζητούν έναν πιο ε, νομικά δεσμευτικό κανονισμό σε σχέση με αυτό που επιθυμούν τα μέλη της, της Επιτροπής. Η θέση μας είναι, θα έλεγα, ρεαλιστική. θα φτάσουμε μέχρι το σημείο που θεωρούμε ρεαλιστικό. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε ήδη σε αυτό το σημείο της έκδοσης σύστασης προς τα κράτη-μέλη για το θέμα ε, της ρύθμισης των συλλογικών αγωγών και αποζημιώσεων στη δική τους ένωμη τάξη και στο δικό τους δικαστικό σύστημα. Ε, εξάλλου, ε, αυτή η έννοια της συλλογική αγωγής και αποζημίωσης απορρέει από εθνικές ενόμες τάξεις κάποιων κρατών μελών. Θέλουμε το νέο εργαλείο να είναι όσο κρατεότερο γίνεται και θα θέλαμε η Επιτροπή να συνεργαστεί στενά ε, με τα κράτη-μέλη ώστε οι συστάσεις που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμοστούν στο μέγιστο δυνατό αριθμό κρατών μελών ενεργειακές τιμές και ε, τιμές ενέργειας μάλλον και αυτά ωφέλη που μπορεί να προκύψουν από ανάληψη λογικής δράσης σε αυτό το τομέα. Το τρίτο πακέτο, το τρίτο ενεργειακό πακέτο φέρνει ε, μεγαλύτερη απελευθέρωση στον ενεργειακό τομέα, επισύρει, επιφέρει μάλλον χαμηλότερες τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια και για το φυσικό αέριο. Και αυτό που θέλει τώρα η Επιτροπή είναι να ενισχύσει περισσότερο τις διατάξεις στον τομέα της τιμολόγησης, ώστε οι λογαριασμοί να είναι σαφέστεροι, πιο διαφανείς, πιο ευανάγνωστοι για τους καταναλωτές. Αυτή είναι μία γραμμή δράσης. Άλλη σχετίζεται με την αρρωγή προς τους καταναλωτές ώστε να εξοικονομούν την ενέργεια. Αυτό συνδέεται φυσικά και με την γραμμή μας για τιμολόγηση. Και η τρίτη γραμμή δράσης είναι διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου. Σε κάποια κράτη-μέλη αναπτύχθηκαν συστήματα συλλογικής ε, μεταφοράς από μία εταιρεία στην άλλη για την παροχή ηλεκτρικής ε, ενέργειας ή φυσικού αερίου. Εμείς θέλουμε να επεκταθεί και να διαδοθεί αυτή η πρακτική και σε άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Συναλόβα έχει ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν συνέχεια να μιλήσουν για να συγκεντρώσουμε όλα τα αιτήματα ώστε να έχει χρόνο ο Επίτροπος να απαντήσει σε όλους. Παρακαλούμε κυρία Συνάλλομο. Eh, Καλησπέρα, κύριε Επίτροπε, και να ζητήσω συγγνώμη από ορισμένους συναδέλφους που είχαν έρθει στην ώρα τους. Ε, ε, εγώ καθυστέρησα γιατί ήμουν αναγκασμένη να παραβρίσκομαι σε άλλη επιτροπή. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, κύριε Επιτροπέ, σε μια προβολή ε, της τσεχικής ταινία που προβλήθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Και συζητήσαμε το ζήτημα της υλοποίησης και της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας. Μετά από πέντε χρόνια από την υιοθέτηση της οδηγίας για τις αθέμητες πρακτικές, η κατάσταση δεν έχει δεν έχει αλλάξει, συγγνώμη. Επομένω, καλωσορίζω την δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσετε στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Το Μάρτιο του 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναφέρει ότι θα εστιάσει περισσότερο στην συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών στα κράτη-μέλη. γιατί εκεί που μετέρχονται θέμη των πρακτικών είναι ιδιαίτερα εμφάνταστοι και βρίσκουν νέα κόλπα κάθε φορά. Με το που θα ξεκινήσει η αντιμετώπιση, η καταπολέμηση μιας αθέμετης πρακτικής, οι εταιρείε αυτές βρίσκουν μια καινούρια ή μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους προς άλλες χώρες. Επομένω, χρειάζεται συνεργασία, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Και το ερώτημα μου τώρα, ε, μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση είχε ανακοινωθεί το 2013 το, με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών. Αλλά προσωπικά δεν διαπίστωσα κάποιες δραστηριότητες ε, αρκετά σημαντικές οι ορατές στον τομέα αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω τι είδους ε, δραστηριότητες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή για την ε, ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Και η δεύτερη μου ε, ερώτηση έχει σχέση με τις αθέμητες πρακτικές και συγκεκριμένα όταν κάποιες εταιρείες οργανώνουν ε, συστηματικά κάποια παρουσίαση για να δελεάσουν τους καταναλωτές. Κύριε Επιτρόπε, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω. Το... Εκτιμούμε ότι επικοινωνείτε και συζητάτε με την Επιτροπή μας τακτικά και μακάρι αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον θα ήταν χρήσιμο. Διάφορα ζητήματα θα ήθελα να ε, συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω με το ζήτημα της επίλυσης συγκρούσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εργαστήκαμε πολύ καιρό για να καταλήξουμε στην τελική οδηγία. Και στην διάρκεια αυτής της προσπάθειας υπήρξαν προβλήματα. Αναφερθήκατε στον ρεαλισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εγώ θα ήθελα να πω να επισημάνω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν ήταν καθόλου ρεαλιστική. Εμείς την κάναμε ρεαλιστική τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να με ενημερώσετε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό. Πώς εκτιμάτε την μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο αυτή τη οδηγία από τα κράτη-μέλη. Ίσως κάποια κράτη-μέλη να χρειάζονται υποστήριξη ή συντονισμό, έτσι ώστε το σύστημα ADR να μεταγραφεί με τέτοιον τρόπο που να είναι συνεκτικό ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Υπάρχουν επίσης προβλήματα χρηματοδότηση αυτού του εγχειρήματο. Διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε του απαιτούμενου πόρου, για παράδειγμα, να ε, χρηματοδοτήσει το σύστημα μετάφρασης που είναι απαραίτητο για ένα online σύστημα επίλυσης συγκρούσεων. Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν ε, επιλύσατε αυτό το πρόβλημα, αν επιλύσατε το πρόβλημα της μετάφρασης και ίσως να ήταν σκόπιμο κάποια στιγμή να παρουσιάσετε, να έρθετε να κάνετε μια παρουσίαση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Είναι ένα ζήτημα που το θεωρούμε σημαντικό και ε, έχουν ανακύψει πολλά ερωτήματα από τους πολίτες. Μια και έχω λοιπόν το λόγο, θα ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία Γκέπχαρτ για το ζήτημα της χώρας προέλευσης, το Made in. Ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οργανώσεις καταναλωτών έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και με ενημερώνουν ότι οι πληροφορίες προέλευσης είναι στην πραγματικότητα παραπλανητικές, γιατί πολλά προϊόντα κατασκευάζονται σε πολλές διαφορετικές χώρες. Η γερμανική λύση, δηλαδή το γεγονό ότι ε, η παροχή αυτών των στοιχείων γίνεται σε εθελοντική βάση, δίνει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στους ε, κατασκευαστές, αλλά τουλάχιστον δεν είναι παραπλανητική προς τους καταναλωτές. Αυτή λοιπόν η λύση που χρησιμοποιείται στη Γερμανία, η εθελοντική αναγραφή, η εθελοντική ενημέρωση, είναι η καλύτερη δυνατή, γιατί αποφεύγει την παραπλάνηση των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Η Μαρία Πέρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Θα επανέλθω λίγο σε ένα από τα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα που είναι το δικαίωμα στην υγεία και σε μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς συγκριτικά μειονεκτήματα ή ε, κοινωνική ανισότητα. Τα πιο καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι και τα πιο ακριβά. Όταν μιλούμε όμως για ισότητα και δεν σκεφτόμαστε τα κοινωνικά δικαιώματα, αυτό είναι εις βάρος της Ευρώπης και την απαξιώνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα απαντήσει στις επιθέσεις που υφίστανται οι Ευρωπαίοι. Στη χώρα μου από αύριο αυξάνεται η συμμετοχή ε, των ασθενών και μπαίνει εισιτήριο στα νοσοκομεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μετσόλα. Grazzi, eh, mistoqsija hija ispirata minn waħda li għadha kif għamlet il-kollega tiegħi. Ευχαριστώ. Ε, με ενέπνευσαν προηγούμενες ερωτήσεις για να επιμείνω κι εγώ για αυτήν την ε, επιγραμμική επίλυση διαφορών, ODR. Στα πλαίσια του, της πρότασης που έχει γίνει το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες για το μεταφραστικό εργαλείο και ξέρουμε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως από ε, το πρόγραμμα διότι έχει περικοπεί ο συνολικός ε, προϋπολογισμός. Θα ήθελα να μας πείτε αν εξακολουθείτε ε, να τηρείτε τη δέσμευσή σας ε, ε, για τη μετάφραση, για τα μεταφραστικά ζητήματα. Ασχολείστε με το θέμα της χρηματοδότησης. θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο που θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα που έθεσαν υπόψη μας ε, τα μέλη της Επιτροπής. Για τις αθέμητες πρακτικές που με τόσο τραγικό τρόπο αποκαλύφθηκαν και αυτή η εταιρεία. Ήταν το αντικείμενο της ταινία που προβλήθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο. πρόκειται για αθέμητες πρακτικές που υφίστανται οι ηλικιωμένοι. Όταν ε, θα απαντούσα ότι φυσικά η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη, τη προστασία των καταναλωτών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό και άρα καλύτερη συνεργασία των αρμοδίων εθνικών αρχών για ευρέως χρησιμοποιούμενες ε, καταχρηστικές αθέμητες πρακτικές. Στη δημόσια διαβούλευση για τη συνεργασία για τα θέματα προστασίας των καταναλωτών ανάμεσα στις εθνικές αρμόδιες αρχές είναι ένα σημαντικό βήμα για να το επιτύχουμε. Πολύ, συχνά, ε, συγγνώμη, πολύ σύντομα θα δρομολογηθούν οι διαβουλεύσεις και θα είναι η ευκαιρία για όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές ώστε να αναφέρουν, να εντοπίσουν και να αναφέρουν τις ε, βασικές τέτοιες αθέμητες πρακτικές για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης των και να διαδοθούν στη συνέχεια στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δεν είναι λοιπόν μία απλή ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην Επιτροπή Αφενός και των Αρμοδίων Εθνικών Υπηρεσιών Αφετέρου. Όχι. Εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς εξ αρχής ενώσεις καταναλωτών, Φερρυπίν. Και η έκθεση που θα ε, προκύψει, ε, με ευελπιστώ ότι θα ενισχύσει και την εθνική νομοθεσία. Ε, για την προστασία των καταναλωτών. Οι εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυση των διαφορών συμπεριλαμβανομένου και του επιγραμμικού τρόπου επίλυση διαφορών, ADR και ODR, είναι τα βασικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για να ρυθμίσουμε διαφορές όπου εμπλέκονται καταναλωτές. Φυσικά θέλουμε καταναλωτικά κέντρα, συμβουλευτικά κέντρα για τους καταναλωτές να συστηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μηχανισμοί, οι εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και οι επιγραμμικές πλατφόρμες ODR, χάρη στις οποίες οι καταναλωτές ε, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους στη δική τους γλώσσα και με βοήθεια που όχι μόνο είναι φτηνό, και διαφανέστερη αλλά και αποτελεσματικότερη σε σχέση με μια δικαστική επίλυση αυτών των διαφορών. Επαναλαμβάνω πως οι επιγραμμικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών όπως προβλέπετε και από τον κανονισμό, θα αρχίσουν να λειτουργούν από Πρώτη του 2016. Η Επιτροπή θα προσφέρει όλα τα πετούμενα μέσα οικονομικά, τεχνικά και ούτω καθεξής για να έχουμε την 1η πρώτη 2016 μια επιγραμμική πλατφόρμα που θα λειτουργεί. Ε, η χρηματοδότηση εν μέρη προέρχεται από τα προγράμματα προστασίας των καταναλωτών. Δεν επαρκούν τα κονδύλια Εκ παραλίλου για την επιγραμμική πλατφόρμα θα βρούμε πηγές χρηματοδότησης και τονίζω και πάλι ότι θα λειτουργεί πλήρως αυτή η πλατφόρμα το 2016. Very important uh, uh, question or, or a comment on. Υπήρξε και μία ερώτηση για το σύστημα υγείας και τα προβλήματα που αυξάνονται και δικαίως ε, για, τα, για τη χρηματοδότηση. Ο Επίτροπος Αρμόδης για τα καταναλωτικά ζητήματα θα μπορούσε να παίξει ένα καταλητικό ρόλο σε συνεργασία με άλλους συνορμοδίους επιτρεωβούς για να θέσει αυτά τα ζητήματα να δώσει νέα όθηση και να προστατεύσει ε, τα συμφέροντα των καταναλωτών. Με τον Επίτροπο Μπος θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε με σφαιρικό τρόπο να οργανώσουμε το σύστημα ούτω ώστε οι ασθενείς να μην πληγούν επουδενή από τις, ε, ε, τα χρηματοδοτικά κενά ε, που χαρακτηρίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας σε πολλά κράτη-μέλη. Στον προηγούμενο γύρο ερωτήσεων ε, με ρωτήσατε ε, για το πακέτο ιατροτεχνολογικών προϊόντων ε, τι πιστεύω για την επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια των καταναλωτών και την ανάγκη να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως δε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αυτές οι ΜΜΕ, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο ήδη ε, στην παραγωγή καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί η ισορροπία, αλλά Το πακέτο ως έχει τώρα προέκυψε από τις προτάσεις Επιτροπής ε, όπως τροποποιήθηκαν από το Κοινοβούλιο συγκλίνει προς μία ενιαία κατεύθυνση. Το πακέτο αυτό σίγουρα δεν θα θέσει εν κινδύνο την ασφάλεια των προϊόντων ή των καταναλωτών και ταυτόχρονα, όπως σας έλεγα, η των καταλλωτων και ταυτοχρονα οπως βιομηχανία θα παραμείνει στην εχμή της τεχνολογίας. Ε, τα συστήματα αδειοδότησης ε, προθέσεις εμπορία των νέων καινοτόμων ιατροτεχνολογικών ε, συσκευών μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε αυτήν την ε, θέση στην αιχμή της τεχνολογίας που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τις ε, απαντήσεις σας, ε, Επίτροπο. Θα μας δοθεί και πάλι ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα που είναι δική σας αρμοδιότητας, αλλά και τα ζητήματα που αποσχολούν και συναρμοδίους επιτρόπους και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ σας ευχαριστώ. Και τώρα θα διακόψω τις εργασίες μας μέχρι τις 5... 4 και 10. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που είναι σε άλλες επιτροπές, πρέπει όμως να έρθουν να ψηφίσουν. 10 λεπτά και διακοπή ακριβώς. Πολύ σας ευχαριστώ. Εγώ το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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να καθίσετε, μπορούμε να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε Σουηδούς προσκεκλημένους και τους καλωσορίζουμε. Αν έχετε την υπομονή να περιμένετε να παρακολουθήσετε τις ψηφοφορίες μετά τις ψηφοφορίες, αλλά μόνο μετά τις ψηφοφορίες, ε, ε, μπορούμε να σας αφήσουμε να καθίσετε. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον την πρώτη ψηφοφορία να την κάνουμε και μετά θα σας καλωσορίσουμε. Σε l'onorevole prende posto. Αν θέλει να καθίσει ο κύριος Ταραμπέλα, αξιότιμος βουλευτής. Allora. Λοιπόν, ψηφοφορία πρώτη έγκριση του χρονοδιαγράμματος για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας για το έτος 2014. Σας έχει διανεμηθεί, έχει εγκριθεί και από τους συντονιστάς και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επικυρώσουμε πλέον το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως το προτείνουν οι συντονιστές μας. Συμφωνείτε? Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Εάν συμφωνείτε με το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής ΙΜΚΟ για το 2014. Va bene. Il Καλώς. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Τώρα μπορούν οι προσκεκλημένοι μας με την ησυχία τους να καθίσουν και εμείς να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μετά, επόμενη ψηφοφορία είναι η έκθεση της κυρίας Μαρίας Ριγκόιεν Πέρες για την ηλεκτρονική υγεία 2014-2020. Έχετε τους καταλόγους σας. Πάμε λοιπόν. Ψηφίζουμε. Η τροπολογία υπαριθμών 1. Παρβανόβα. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Η κοντράρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2. Προσθήκη της κυρίας Λεγκρίπ. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Voto è aperto. Αρχίζει η ψηφοφορία. Il voto è chiuso. È approvato. Ε, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. θα σας παρακαλούσα να, χρειάζεται τα χέρια, να σηκώνετε τα χέρια σας για να σας βλέπω. Να μην κάνουμε συνέχεια ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ε, δεν μπορώ πάντα να βλέπω τι ψηφίζει, δεν είναι δύσκολο. Τρία, ποιοτικά είναι ψηφί παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τοπολογία 4, Ποιετικά είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 ε, της εισηγήτριας είπε κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. il voto. Άρχεται πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Πιετικά είναι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία τώρα 13 και 14 μου είναι με συμπράσεις και πάξας. Ηλεκτρονικά κατευθείαν αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απροβάτο. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 ψήφι Πέρα παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Παρβάνοβα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22-23. Εμβράσας και Ρολάνδας. Πάξας. Αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 τροπολογία. Ποιοτικά είναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 Παρβάνοβα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 Παρβάνοβα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 6 υπέρ συμβαστική κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε τώρα το σύνολο ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχιτε ψηφοφορία Πέρασε. Relazione approvata, 30 voti. 30 υπέρ και μία ψήφο ε, κατά. Συγχαρητήρια κυρία Ριγκόγεν. La relazione successiva. Επόμενη έκθεση. είναι της κυρίας ε, Γκάλ Πέλτς. για ε, την τεχνολογική και βιομηχανική βάση στην Ευρώπη για την αμυντική βιομηχανία. Έχετε τον κατάλογο σας. Ε, πάμε. Ε, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 4. Όχι. Η δύο έχει καταπέσει. Η τέσσερα. Γκέπχαρτ. Υπέρ. Τέσσερα, η είναι της κυρίας Γκέπχαρτ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δύο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική τρία κατά τμήματα. Πρίμα πάρτε. Τμήμα πρώτο. Κύριε Γκέπχαρτ, διαπιστώνω ότι δεν έχω υπογράψει αυτή τη συμβαστική τροπολογία όπως λανθασμένα αναφέρει ο κατάλογος ψηφοφορίας. Okay. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε ψηφίζουμε κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον του συμβαστικού τρία, Τμήμα, ε, υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεν κρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ψήφι κατά, απόχες, εγκρίνεται, 15, χάρπορ, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 16 όλες μύτη υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 17. Γκέπχαρτ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 19 Σφαμπ. είπε, Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 20 Γκάλπελτ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 Σμιτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 Βάιλερ υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 23, 24, 25 μαζί να τις ψηφίσουμε, συμφωνείτε, Όμπερ Μάιερ, υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτονται, συμβαστική 4, υπέρ, κατά, άποχες, α, εγκρίνεται, 29, της ιδέας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 30 Γκέπχαρτ είπε. κατά αποχές εγκρίνεται 31 Μπιέλαν είπε. κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ αρχίζει τώρα η ψηφοφορία Πέρασε. Εγκρίνεται. 32 Γκέπχαρτ είπε Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 33 Μπιέλαν υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Πέρας. Approvato con 19 voti a favore. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 11 κατά, ε, χωρίς αποχ... Ε, δύο αποχές, συγγνώμη. Bene. A questo punto abbiamo finito la parte relativa. Τελειώσαμε εδώ λοιπόν ε, τις ψηφοφορίες. Δύο λεπτάκια να δώσουμε στους συναδέλφους που θέλουν να αποχωρήσουν οι ανυποχρεωμένοι γιατί έχουν άλλες ανηλυμένε υποχρεώσεις και μετά θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Δύο λεπτά ακριβώς το διάλειμμα. giustissimi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 Bene, possiamo riprendere Πέρασαν είναι τα δύο λεπτά και πρέπει εγώ να κάνω την παρουσίαση για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μου έχει ανατεθεί αυτή η έκθεση. Ε, είναι η πρώτη συζήτηση που κάνουμε για αυτήν την έκθεση. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στην ανακοίνωσή της Ήταν μια ανακοίνωση που σχετιζόταν άμεσα με τις δικές μας εργασίες, διακυβέρνηση δηλαδή, στον τομέα της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο ότι Παρότι η εμέ είναι πάρα πολύ σημαντική η ενιαία αγορά, το θέμα τώρα είναι να ε, είμαστε σε επαγρύπνηση ούτως ώστε να υπάρχουν οι απαιτούμενες διαδικασίες ενισχύ ούτως ώστε στο μέλλον, στα πλαίσια της ετήσιας ε, ανάλυσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να υπάρχει μια ειδική έκθεση για τα ε, πεπραγμένα στην ενιαία αγορά, για το στάδιο ολοκλήρωσής της. Ε, στη συνέχεια, έχουμε την έκθεση ΣΦΑ που έχει ψηφιστεί ψηφίστηκε στην ε, Ολομέλεια μαζί με άλλες εκθέσεις που σχετιζόντουσαν ε, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ενισχύουμε λοιπόν τη θέση μας και το ρόλο της Επιτροπής μας σε σχέση με το παρελθόν. Όπως γνωρίζετε, ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώνει κατά πόσο ε, υλοποιείται από τα κράτη-μέλη η στρατηγική 2020. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να περιορίζουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους σημαντικούς πυλώνες της ε, οικονομικής, πολιτικής ε, αφενός και της κοινωνικής πολιτικής αφετέρου, διότι είναι αλληλένδετοι αυτοί οι δύο πυλώνες ως προς την κείμενη νομοθεσία και ως προς ε, τη λειτουργία της ενίας αγοράς. Αυτό το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς μπορεί να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες ε, της Επιτροπής και ε, προσδίδει ένα πολιτικό περιεχόμενο μέσα από τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι επακριβή μεθοδολογία συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ούτως ώστε να κατοχυρώνουμε την ε, ολοκλήρωση αυτών των τριών πυλώνων ε, και να επιτύχουμε ώστε να επικρατήσουν κοινέ αξίε. Έχουμε τομεί κλειδιά που αναφέρονται στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θυμάστε ότι πρόκειται για τις υπηρεσίες, στη συνέχεια χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίες, μεταφορές, ενέργεια και ε, ψηφιακή ενιαία αγορά. Εγώ κρίνω πως θα ήταν χρήσιμο να προσθέσουμε επιπρόσθετα ζητήματα αξιολόγησης που θα σχετίζονται πιο συγκεκριμένα με την ε, προστασία των συμφερόντων των ε, καταναλωτών διότι ε, οι καταναλωτές με τις διαφορετικές ιδιότητες που έχουν, οικονομικοί φορείς δηλαδή οι καταναλωτές, μετέχουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να προσδώσουμε την δέουσα σημασία στους ε, καταναλωτές. Είναι εξάλλου αυτοί που μας ψηφίζουν, οπότε ε, θα πρέπει να προστατεύουμε τα συμφέροντά τους σε ε, ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Η έκθεση ΣΦΑΠ βασιζόταν Ε, στην πράξη για την ενιαία αγορά και στη δεύτερη εκδοχή αυτής που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή όταν εμείς ψηφίζαμε την έκθεση σβαπ Τώρα μπορούμε να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο αυτής της νομοθετικής πράξης έχοντας ε, καλύτερη επίγνωση της πραγματικότητας. Η έκθεσή μου θα αναλύσει επίσης τα εργαλεία χάρη στα οποία θα προσδιορίσουμε επακριβέστερα την ενιαία αγορά, αξιοποιώντα παλαιότερα εργαλεία και θεσπίζοντας νέους ελέγχους και επαληθεύσεις που θα είναι τέτοια ώστε να λαμβάνονται υπόψη ε, τα συμφέροντα των καταναλωτών. Δεν θα αξιολογήσουμε μόνο ποσοτικά ή ποιοτικά ε, πρότυπα, θα εισακουστεί η φωνή των καταναλωτών για τις επιμέρους δράσεις αλλά και για το περιεχόμενο της ε, ενιαίας αγοράς. Αυτά είναι τα βασικά σημεία αναφοράς, διότι αυτά είναι και ε, αυτά, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν ε, καθημερινά εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, στις 15 Οκτωβρίου θα καταθέσω την έκθεσή μου, θα έχετε και χρόνο για να συζητήσουμε την έκθεση. Η καταληκτική ημερομηνία που έχει προβλεφθεί προς το παρόν για τις τροπολογίες είναι 15 Νοεμβρίου. Ε, προβλέπεται προς το παρόν, λέω, διότι αν στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταθέσει την ε, ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, ε, τότε ε, θα χρειαστεί να αναβάλουμε την καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτού καταθέσουν τις τροπολογίες τους. Προς το παρόν λοιπόν 15 Οκτωβρίου παρουσίαση, 15 Νοεμβρίου οι τροπολογίες, παρακαλώ και το τονίζω, ενδέχεται να τροποποιηθεί αυτή η ημερομηνία ε, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάξει το χρονοδιάγραμμά της ε, για την πρότασή της. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αν δεν αλλάξει τίποτα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες, θα περάσουμε μετά στις συμβαστικές τροπολογίες. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στους κοιόδης από τις διάφορες πολιτικές ομάδες που έχουν ε, δηλώσει την επιθυμία τους να μιλήσουν. Άνσλικ από το ΕΛΚ. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałabym się wypowiedzieć również w imieniu pana e, Andreasa Schwaba, koordynatora IPP e i sprawa... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντρέα Σβάπ ε, που είναι ο συντονιστής του ΕΛΚΑ και έχει αναλάβει την έκθεση για την ενιαία αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ενιαίας αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια έκθεση για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να ε, κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, για αυτή την έκθεση ΣΒΑΒ. Πρώτον, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως οι αρχές της ενιαίας αγοράς μετά από την αξιολόγηση που θα γίνει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δυστυχώς δεν <clears throat> υπάρχει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Είναι Παρότι δεν είναι παγιωμένο, όπως θα θέλαμε η νέα αγορά, είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε τις αρχές της, να προωθούμε κυρίως τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, γιατί αυτό θα επιτρέψει δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τονίζει ο κύριος Φαπ ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι σημαντικό οι δικές συστάσεις αναχώρα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρώνονται περισσότερο ε, στις ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο στην εφαρμογή αυτών των ειδικών συστάσεων και αντί να χάνουν το χρόνο τους απορρίπτοντας αυτές τις συστάσεις όπως έκανε η Γαλλία. Κάποιες από τις προτάσεις του κυρίου Σβάπ έχουμε ήδη εφαρμόσει ενισχυμένη χρήση νέων εργαλείων για την ε, συλλογή δεδομένων και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια σχετική έκθεση ε, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες σε ένα επικοδομητικό πνεύμα και προσβλέπουμε στη μελλοντική μας συνεργασία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριο Χατζημαρκάκη από του Φιλελευθέρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν τη σημασία αυτής της έκθεσης με εξαίρεση εκείνους που ασχολούνται με το θέμα. Πριν από τρία χρόνια είδαμε το θέμα του ε, κρατικού χρέους και της κρίσης και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ωραία όλα αυτά, αλλά ξεχάσαμε ότι όλοι οι παράγοντες που οδηγούν στην υπερχέωση των κρατών, δηλαδή μείωση της παραγωγής, μείωση της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξη σε κάποια χώρα, οδηγεί σε μεγαλύτερη χρέωση και αυτό έχει πολύ μεγάλη θέση με την ιστορική αγορά. Οπότε είναι απολύτω λογικό Κανονικά θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα θέματα αυτά της οικονομικής ανάπτυξης, ε, της υπόθεσης του χρέους, να τα βλέπουμε και από το πρίσμα και ε, σε συνδυασμό με την εσωτερική αγορά. Όπως είπε πολύ ωραία στην έκθεση του ο κύριος Φαμπ, βεβαίως πρόκειται για την εφαρμογή, αλλά όχι μόνο για την εφαρμογή. 20 χρόνια κλείνει, έκλεισε η ε, εσωτερική αγορά και 10 χρόνια η ΟΝΕ και δεν είναι μόνο η εφαρμογή αλλά είναι και συμψηφισμός και ε, μη Εγώ έχω επικότητα σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τα δύο άκρα αν θέλετε. Στην τελευταία τριετία ε, η μία μου πατρίδα, η Ελλάδα, έχασε ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, ενώ η άλλη μου χώρα που την ξέρω πολύ καλά, η Γερμανία, δημιούργησε ένα μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μπορεί προσωρινά να είναι βιώσιμη, αλλά εις το διηνεκές είναι αφόρητη. Εμείς ως Ευρωπαίοι λοιπόν πώς ε, θα το αξιολογήσουμε αυτό. Έχουμε ένα βαθμολόγιο, ένα scoreboard λεγόμενο, το τελευταίο πότε ήτανε. 19 Φλεβάρι του 2013 λέει εδώ και διαπιστώνουμε ότι σε αυτό το βαθμολόγιο κάποιες αρνητικές επιπτώσεις όπως είναι επιθετική πολιτική εξαγωγών στην εσωτερική αγορά ε, ε, ε, μπορεί να έχει την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον, συγγνώμη, να τις επιπλήττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά στη Γαλλία που την επέπληξαν δεν το έλαβε και πολύ υπόψη της. Η Γερμανία το βλέπει θετικά γιατί έχει πλεόνασμα και μεγάλο και απλούστατα ε, τις αγνοεί αυτές τις επιπλήξεις η Γερμανία. Και κάποιος συνάδελφος, κάποια συνάδελφος προηγουμένως είπε ότι ε, ό,τι ισχύει για τη Γαλλία ισχύει και για τη Γερμανία. Ναι, αλλά κάνει συστάσεις χώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εάν κανείς δεν τις λαμβάνει υπόψη, τις αγνοεί απλούστατα, τότε μπορούμε να το κλείσουμε το μαγαζί και θα δούμε ότι η εργασία θα συγκεντρώνεται στο γεωγραφικό κέντρο της Ευρώπης και η περιφέρεια θα τονίζει και θα ε, λησμονείται. Σε χώρες λοιπόν που έχουν πλέον άσματα θα πρέπει πραγματικά να επιδοτούν τον κόσμο για να πηγαίνουν διακοπές στις χώρες του Νότου. Ξέρω εγώ, οικονομικά αυτά που σας λέω βγαίνουν. Αν το πω πολιτικά στη Γερμανία, νομίζω θα με πετάγαν έξω από την αίθουσα και θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό ε, με συνέπεια. Ο κύριε Κοφεράτη, κύριε ε, Πρόεδρε, η έκθεση αυτή είναι μια δυνατότητα να κάνουμε τη φωνή του Κοινοβουλίου να ακουστεί, γιατί θα πρέπει να φωνάξουμε ξανά, αλλά τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, υλοποιούν τα όσα γράφουν, γιατί πραγματικά είναι διασπάθηση των χρημάτων των φορολογουμένων και καταστροφή θέσεων εργασίας σε κάποιες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Αν όχι, θα παρακαλούσα τους κυρίους που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θέλουν να ε, σχολιάσουν τα όσα άκουσαν. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς. Θα μου ξαναδώσω το λόγο <laughs> για να πω κάτι πάρα πολύ σύντομα. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο. Το πραγματικό πρόβλημα ποιο είναι. Θα πρέπει να δώσουμε νόημα σε αυτό το τρίτο πυλώνα που είναι η ιστορική αγορά. Το Κοινοβούλιο θεωρητικά και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως και το Συμβούλιο Σημερίζονται αυτές τις απαιτήσει, αλλά στην πράξη διαφέρουν πάρα πολύ τα πράγματα. Καμία σχέση με ε, τις ε, θεωρητικές μας τοποθετήσεις. Εμείς θα πρέπει να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα, αυτή τη διαφορά, αυτή είναι η δουλειά μας. Να κάνουμε εφαρμόσιμα και υλοποιήσιμα αυτά τα περιεχόμενα της έκθεσης ΦΑΠ και να ενισχύσουμε ακριβώς το ευρωπαϊκό εξάμεινο και να υπάρχει μια διασύνδεση, μίας ένας συσχετισμός ανάμεσα στις οικονομικές πολιτικές, στις κοινωνικές πολιτικές και στις πολιτικές της εσωτερικής αγοράς. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ελέγχουμε, θα το κάνουμε και θέλω να θυμίσω σχετικά ότι, όπως σας είχα πει, οι προθεσμίες που ισχύουν είναι εξής. 15 Οκτωβρίου θα έχετε την έκθεση και στις 15 Νοεμβρίου, εάν δεν υπάρξει κανένα πρόβλημα από την Επιτροπή, έχετε την προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών σας. Τούτο λεχθέντων, παίρνουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης και θα δώσω και πάλι στον εαυτό μου το λόγο Είναι μια γνωμοδότηση ε, που είμαι εγώ συντάκτης με θέμα την αποκάλυψη προφοριών μη οικονομικής φύσεως οδηγία είναι και προφοριών σχετικά με την πολυμορφία σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι αυτές. Επί τη ουσία αρμόδια είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, εμείς γνωμοδοτούμε. Πώς γεννιέται αυτή η οδηγία delle due opinioni είχαν εγκριθεί δύο οδηγίε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και έχουμε στα χέρια μας επίσης και το έγγραφο της Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης λαμβάνονται μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα. Αυτό έχει προχωρήσει αρκετά στην Ευρώπη. Μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια από τι σημαντικότερε καινοτομίε που εισήγαγε η Λευκή Βίβλο του Ζακ Τελόρ το 1993 ήδη. Αυτέ οι πρακτικέ σιγά σιγά υιοθετήθηκαν από όλο και περισσότερου μετά από δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη επιτροπή του Κοινοβουλίου, αλλά παραμένουν ε, μέτρα εθελοντικά. Και το κεντρικό στοιχείο ε, κίνητρο για την ανάληψη πρωτοβουλειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι η φήμη μιας εταιρείας. Έχουν υπάρξει και κάποιες ε, οπισθοχωρήσεις και κάποια πισωγυρίσματα, κάποια στοιχεία τα οποία δεν υλοποιήθηκαν. Αλλά και μεγάλες αντιφάσεις ανάμεσα σε εκείνες τις πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καταπτύσσουν υπέροχες εντυπωσιακέ εκθέσεις για την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη τους και τα προγράμματά τους που τα παρουσιάζουν όλα υπέροχα και εξοραϊσμένα αλλά ανάμεσα σε αυτές τις εταιρείε μπορεί να είναι για παράδειγμα οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείε, οι οποίες ενώ μας παρουσιάζουν τρομερά προγράμματα κοινωνική ευθύνη, ευθύνονται για τις πετρελαιοκυλίδες στη Βόρεια Θάλασσα. Εξαιτία τη ε, πρακτική του να μεταφέρουν το πετρέλαιο με ε, τάνκερ που δεν ε, πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας ή επίσης μπορεί να πρόκειται για εταιρείε που εκμεταλλεύονται την παιδική εργασία στην Ασία. Και συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολο να αναγκάσουμε αυτές τις εταιρείες να ακολουθήσουν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η επισης μπορει να προκειται για εταιρειες που εκμεταλλευονται την παιδικη εργασια παρέλαβε τις δύο ε, γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τις προτάσεις της Επιτροπής. Θα έλεγα ότι είναι καλά δομημένη και με καλές προθέσεις η πρόταση της Επιτροπής. Αυτό που θα έπρεπε εμείς πιστεύω να κάνουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου είναι να αυξήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τη διαφάνεια, κάτι που θα ευνοήσει τους πάντες και ιδίω του καταναλωτέ, που είναι οι, ε, εκείνοι που ενδιαφέρονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για να γνωρίζουν τις πραγματικές δραστηριότητες μιας εταιρεία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αλλαγές που θα μπορούσαμε να κάνουμε διατηρώντας τη δομή του κειμένου ως έχει. Γι' αυτό έχω υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες. τροπολογίες αυτές θα πρέπει να είναι να συνάδουν με την πρωτοβολία που είχε αναλάβει το Κοινοβουλίο από την αρχή. Λοιπόν, για το ζήτημα του κατοφλίου, ε, με βάση το οποίο θα ε, επιλέγονται οι μεγάλες εταιρείες, η Επιτροπή προτείνει τους 500 εργαζόμενους. Εγώ προτείνω 250. Γιατί ε, με αυτό το κατόφλι καθορίζονται οι μεγάλες εταιρείες σε όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 250 εργαζόμενοι δύσκολα θα μπορούσε ο να επιχειρηματολογήσει, γιατί στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να έχουμε άλλο κατόφλι. Και όχι τους 250 εργαζόμενους που χρησιμοποιούμε και επιβάλλουμε σε όλα τα άλλα νομοθετήματα. Επίσης θα έπρεπε να διευκρινιστεί η έννοια του κινδύνου. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να είναι ε, όσο δυνατόν πιο ομοιόμορφες οι πληροφορίες που θα παρέχουν οι επιχειρήσεις. Στην πρόσφατη συζήτηση που είχαμε για τις δημόσιες ε, προμήθειες, είπαμε ότι θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να έχουμε την κατάσταση στην οποία μια εταιρεία ε, η ίδια να έχει μια καλή εικόνα όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη, αλλά να μην ελέγχει τους προμηθευτές της και οι... σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η αλυσίδα των προμηθευτών μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη. Χρειάζονται λοιπόν μηχανισμοί ελέγχου. Επαναλαμβάνω ότι δεν αναφερόμαστε σε νομικά δεσμευτικά μέτρα, αλλά εάν μια εταιρεία αρνηθεί να παράσχει αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να το αιτιολογήσει, να εξηγήσει γιατί. Και εν τέλει να ε, αιτιολογήσει αυτήν την επιλογή στους καταναλωτές και στους μετόχους της. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο να βελτιωθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη στα χαρτιά, πρέπει να πραγματώσουμε αυτό για το οποίο συζητάμε ήδη από το 2000 και το οποίο φαίνεται να έχει μείνει πίσω. Με τις πρόσφατες εξελίξεις έχασε κάπως την ε, σημασία που του δίναμε παλαιότερα η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Λοιπόν, με, με χαρά θα ακούσω τις δικές σας προτάσεις ε, και σχόλια, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής. έτσι ώστε να συνάδει και με τα διάφορα άλλα μέτρα που έχει υπερψηφίσει το Κοινοβούλιο στον τομέα της ε, εταιρική κοινωνικής ευθύνης στο παρελθόν. Ε, πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ας μην παραμείνουμε σε μια μειοπική προσέγγιση και απλώς ε, σε μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση. 15 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στη συζήτηση και θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στους Σκιώδης, εισηγητές. Κυρία Πιετικάινεν για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με συγχωρέσετε γιατί τα σχόλια που θα κάνω ε, έχουν επηρεαστεί πολύ περισσότερο από τις προσωπικές μου εμπειρίες παρά από το πολιτικό μου υποβαθρό γιατί έχω μια, επιχείρηση, ε, έχω μια εμπειρία στην διοίκηση επιχειρήσεων και αυτό μου δίνει κάποιες ε, δυνατότητες, κάποιες εμπειρίες, κάποιες γνώσεις που δεν μπορώ να μην λάβω υπόψη μου. Πρώτα λοιπόν, νομίζω ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έως τώρα είναι πολύ θετικό. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, είναι λογικό να επιδιώξουμε να υπάρξει ισότιμο ανταγωνισμό, ισότιμο πεδίο και άρα να απαιτούμε το ίδιο επίπεδο ε, πληροφόρησης από όλες τις επιχειρήσεις του ίδιου μεγέθους. Αυτό μου φαίνεται λογικό. Νομίζω υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που λείπει και στη γνωμοδότηση του εισηγητή και στην πρόταση της Επιτροπής και αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, ποιο είναι αυτό λοιπόν. φανταστείτε την κατάσταση κατά την οποία έχουμε εθελοντικό χαρακτήρα αυτών των μέτρων και ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά συστήματα ε, αναφορών, ε, ενημέρωσης. Αν το δούμε από την πλευρά των επιχειρήσεων, είναι κρίσιμη σημασία στα στοιχεία αυτά να είναι συγκρίσιμα. Γι' αυτό, για παράδειγμα, υπάρχει η οδηγία περιλογιστικών καταστάσεων ή το IFRS, τα, τα, λογιστικά πρότυπα. Φανταστείτε τα λογιστικά πρότυπα να ήταν διαφορετικά και να μην μπορούσαν να συγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις μεταξύ των ε, εταιριών. Ένας επενδυτής ή οποιοδήποτε, εάν δεν μπορούσε να έχει συγκρίσιμα στοιχεία, δεν θα μπορούσε να συγκρίνει δύο εταιρείε και τις ενέργειές τους και τις πολιτικές τους. Τώρα, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, θα έχουμε εθελοντικό χαρακτήρα των στοιχείων. Και η παρουσίαση αυτών των στοιχείων θα γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό οδηγεί σε πλήρη αδυναμία συγκρίσεων. Η κοινή γνώμη είναι πολύ δύσκολο να αποφανθεί Από την πλευρά των επενδυτών επίσης, τη σκοπιά των επενδυτών, στη μία περίπτωση θα, είναι θα, θα, υπάρχουν οι ενοποιημένες καταστάσεις, ε, οι ενοποιημένες συγγνώμη, εκθέσεις και από την άλλη οικονομικές καταστάσεις. Ε, σε ποιες θα βασιστεί ένα επενδυτικό ταμείο, για παράδειγμα, ένα συνταξιοδοτικό επενδυτικό ταμείο, φαντάζομαι στις οικονομικές. Και αυτό ε, ενθαρρύνει μια προσέγγιση του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Μπορεί μια εταιρεία βραχυπρόθεσμα αμέσα να έχει μεγάλα κέρδη, αλλά μακροπρόθεσμα να έχει υποθηκεύσει το μέλλον της. Να μην έχει, για παράδειγμα, επενδύσει επαρκώς στο, στην εταιρική της ταυτότητα ή σε ε, άλλου είδους επενδύσεις. Απ' την άλλη, εάν δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα στοιχεία, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι επενδυτές να μην κάνουν, να μην μπορούν να κάνουν, λέω, την πλέον βιώσιμη αηφόρο επιλογή. Επομένως, στο μέλλον, πέρα από τους κρίσιμους δείκτες τους key performance indicators, θα πρέπει να έχουμε ένα βασικό κοινό σύστημα ε, το οποίο να εφαρμόζεται στις εκθέσεις των εταιριών. Φοβάμαι ότι προχωρώντας έτσι με μικρά βηματάκια, χωρίς να κάνουμε κάτι αποφασιστικό, αυτό που στην πραγματικότητα προκαλούμε είναι απλώς περισσότερη γραφειοκρατία. Απλώς ζητούμε από τις επιχειρήσεις να παράγουν όλο και περισσότερες εκθέσεις και στο τέλος δεν λαμβάνουμε καν τις πληροφορίες που πραγματικά χρειαζόμαστε, που είναι σημαντικές, οι οποίες θα επηρέαζαν τελικά τις επενδυτικές επιλογές. Ούτε υποστηρίζουμε τα μακροπρόθεσμα ε, συγγνώμη, επενδυτικά προγράμματα. Ούτε δημιουργούμε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού. Ε, δεν γνωρίζω ακριβώ θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα άμεσα, γιατί ε, θα, για, να, για ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, θα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση και με τον επιχειρηματικό κόσμο. Επομένως το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή. Αλλά φαντάζομαι ότι τουλάχιστον θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση να συμφωνήσουμε ως προς το πότε θα είναι η ημερομηνία για μια αναθεώρηση που θα οδηγήσει σε κοινού ε, κανόνες για την ε, παροχή αυτών των πληροφοριών, για την, για την κατα... κατάρτιση αυτών των εκθέσεων. Να συμφωνήσουμε μια ημερομηνία σε πέντε χρόνια όπου θα αναθεωρήσουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο και θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Κρόιτσμαν, ο οποίος είναι σκιώδης ηγητής μας. Το θέμα της ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας απασχολεί στο Κοινοβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό τι δείχνει αφενός την ε, αυξανόμενη σημασία αυτών των δραστηριοτήτων των εταιριών αλλά και τη σημασία που δίνει ο κόσμος. Το CSR όπως λέγεται δεν είναι νέο φαινόμενο εδώ και καιρό και πολλές εταιρείες το έχουν υιοθετήσει από παλιά. Η αρχή όμως εδώ είναι η αρχή της ε, ε, Εθελούσια συμμετοχή. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει, αλλά να το αποφασίζει μόνος του ως ελεύθερος επιχειρηματίας. Στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αφιστάμεθα πλέον από την εθελούσια βάση. Είναι λίγο κατασκευασμένη αυτή η πρόταση και ιδεολογικά ε, κινούμενοι. Ειδικά οι εταιρείε που δεν είναι στην ε, προσοχή της κοινή γνώμης, αλλά εκτίθενται ε, στο διεθνή ανταγωνισμό και επιβαρύνονται με επιπλέον γραφειοκρατία και κόστος. Και αποσπώνται από τις βασικές δουλειές τους, που είναι να παράγει κανείς υπηρεσίες ή να κατασκευάζει προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για ε, ε, λίγες εκατοντάδες μέχρι χίλια ευρώ. Αλλά αυτό είναι προβληματικό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε λίγες ώρες να συνοψίσει για τη μελέτη σκοπιμότητας κάποιες εκθέσεις. Μα μπορεί να μην υπάρχει καν ένα αντίστοιχο τμήμα στην εταιρεία αυτή. Τι γίνεται με τις θηγατρικές εταιρείε που θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες ή μάλιστα να ε, αναγκαστούν να συμμετέχουν και εξωτερικοί ελεγκτές. Έρχονται εδώ να προσθεθούν και κάποιες πληροφορίες για την πολιτική διαφοροποίηση και, ε, στις ε, εταιρείε και πολυμορφίες. Ήδη δεν είναι χωρίς πρόβλημα και είναι και πολύ ε, αμφιλεγόμενη η ποσόστοση των γυναικών. Αυτό που θέλουν οι εταιρείε είναι να προσλαμβάνουν τους πιο άξιους. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν τα πάμε καλά στην αγορά επειδή δεν έχουμε αρκετές γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά. Αυτό που ενδιαφέρει μια εταιρεία είναι να έχει τους καλύτερους μάνατζερ με την καλύτερη εμπειρία και την καλύτερη μόρφωση και σπουδές. Πώς μπορούμε εμείς ως νομοθέτες να έχουμε την αξίωση ότι θα παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τις εταιρείες τους από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Αυτό του κυρίου Κρόιτσμαν του φαίνεται περίεργο, ιδιαίτερα και το πεδίο εφαρμογής που ε, επεκτείνεται σε εταιρείε με 250 και πλέον εργαζόμενους. Και μάλιστα ε, είναι επιπλέον το κόστος εδώ εις βάρος άλλων τομέων και είναι και εις βάρος ε, της ανταγωνιστικότητας, ενώ στόχος μας θα πρέπει να είναι ακριβώς το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ δεν βλέπω άλλους κοιόδης. Α, η κυρία Γκέφχαρντ. Παρακαλώ, Εύελιν. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγητά μου. Αγαπητέ Σέρτζιο. Πολύ καλή η έκθεση που προτείνει το σχέδιο και συμφωνώ ε, με την άποψή σας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια καλή καταρχήν πρόταση. Και έχει νόημα πραγματικά αυτή η πληροφόρηση και η διαφάνεια που είναι ε, οπωσδήποτε απαραίτητη να επέρχεται. Και μπορείτε να πείτε στον κύριο Κρόιτσμαν, κύριε Χατζημαρκάκη, αν έχει την καλοσύνη, ότι αν δούμε ποιοι είναι οι κανόνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ποσοστώσεις των φύλων, αυτά εκεί που ισχύουν πολύ πιο αυστηρά από τα όσα ε, περιλαμβάνονται στην πρόταση του κυρίου Κοφεράτη. Οπότε Τώρα να μιλάμε για στρεβλώσεις του ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας στην παγκόσμια αγορά μου φαίνεται κάπως προβληματικό. Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι είναι πλεονέκτημα εάν δημιουργείται τέτοια διαφάνεια και λογοδοσία. Το βλέπουμε αυτό και στην κοινωνία μας όλο και περισσότερο και οι πολίτες και οι καταναλωτές και οι αγοραστές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το τι σημαίνει στα παρασκήνια. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και καλωσορίζω δύο σημεία που ανέφερε ο κύριος Κοφεράτη, δηλαδή συνέπεια στην νομοθεσία και εφαρμογή σε εταιρείε που έχουν από 250 υπαλλήλους και πάνω. Σε πολλές ε, πτυχές και σε πολλά νομοθετήματα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αναφέρεται αυτός ο αριθμός. Είναι από 250 και πάνω. Καλό είναι να υπάρχει μια συνέπεια και να μην επέλθει ένα γενικότερο αλαλούμ. Επίσης αυτό αφορά και κάποιες θηγατρικές. Γιατί τι να την κάνω ε, σε μια μεγάλη επιχείρηση τη διαφάνεια και την ενημέρωση όταν ε, αναθέτουν σε υπεργολάβους διάφορα πράγματα, μόνο θηγατρικές, λοιπόν, θα πρέπει να καλύπτεται και οι υπεργολαβίες εδώ. Είναι δύο σημεία αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και με χαροποιούν στην πρόταση του κυρίου Κοφεράτη. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι. Θέλει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σχολιάσει αυτό το θέμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την έκθεση και για όλες τις διευκρινήσεις που ακούσαμε σήμερα. Τον Απρίλιο ενέκρινε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατά τη γνώμη μας ενισχύει τη διαφάνεια και τις επιδόσεις των, ε, στις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σε σχέση με τις καθημερινές αποφάσεις αλλά και το σχεδιασμό ε, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δράσης των επιχειρήσεων. Αυτό είναι υποφελές και για τις επιχειρήσεις, για να είναι καλύτερες οι αποφάσεις τους, αλλά και για την οικονομική και μη οικονομική βιωσιμότητά τους στο μέλλον. Αυτή είναι η άποψη της Επιτροπής. Αυτή ήταν, ε, αυτό ήταν και το πόρισμα της αξιολόγησης αντικτύπου που κάναμε. Οι επενδυτές και οι ενώσεις τους διαρκώς μας επισημαίνουν πως χρειάζονται τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες για να συμπληρώσουν τις οικονομικές πληροφορίες που ήδη λαμβάνουν. Οι επενδυτές αναφέρουν ότι είναι χρήσιμα αυτές οι πληροφορίες για τις αποφάσεις ε, που, κάνουν, ε, που λαμβάνουν για το κεφάλαιο, παραδείγματος χάρη των επιχειρήσεων, Ε, ε, λαμβάνουν επαρκείς ε, και ποιοτικέ πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία, αλλά όχι για τα μη οικονομικά στοιχεία, όπως έλεγα, για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, που όμως έχουν μεγάλη σημασία για τη λήψη αποφάσεων από πλευρά των επενδυτών. Και θεωρούμε ότι ακολουθούμε τη σωστή προσέγγιση την νομοθετική προσέγγιση. Υπάρχουν 250.000 επιχειρήσεις που είναι ήδη διαφανείς για περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα. Στις αιτήσιες εκθέσεις του συμπεριλαμβάνουν αυτά τα στοιχεία. Εμείς προτείνουμε αυτό το όριο των 500 εργαζομένων και ο αριθμός θα αυξηθεί κατά 600% φτάνοντας τις 18.000 επιχειρήσεις. Ε, είναι μεγάλη πρόκληση για μας, αλλά θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί επιλέξαμε το όριο των 500. Αν είχαμε επιλέξει 250 εργαζόμενους, θα ήταν 45.000 οι επιχειρήσεις που θα στοχεύαμε. Και αναρωτιέμαι αν η αγορά θα άντεχε μια τόσο ριζική αλλαγή. Φυσικά θα μπορούσε αυτό να ε, διευκολυνθεί με νέες τεχνικές ε, ή προσαρμόζοντας τη χρονική περίοδο για τη μεταφορά. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, να μην επιβάλλουμε ένα υπερβολικό άχθος στις επιχειρήσεις. Θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η νέα απέτηση αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή τη χρονική στιγμή δεν θέλουμε να επέμβουμε επιβάλλοντας νέες απαιτήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παραδοσιακό όριο για τις μικρομεσαίες είναι μέχρι τους 250 εργαζομένους. Αλήθεια είναι αυτό όμως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στοχεύσουμε τις πραγματικά ευμεγέθεις επιχειρήσεις. δεν κρίνουμε σκόπιμο να στοχεύσουμε μικρότερες επιχειρήσεις και με αυτό το όριο νομίζω είναι ξεκάθαρο και το μήνυμά μας. Ακούσαμε σχόλια για την παροχή πληροφοριών ε, για όλη την τροφοδοτική αλυσίδα. Είναι απαραίτητο, δεν το αρνούμαστε. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες γιατί είναι χρήσιμες για τις επιχειρήσεις, για τους επενδυτές, για τους μετόχους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιούν τις πληροφορίες για το σεβασμό παραδείγματο χάρη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα βασικότερα ζητήματα με τις υπεργολαβίες είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύουμε ότι το ρυθμίσαμε με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς βεβαίως να ξεχνούμε τις τεχνικές δυσκολίες που δεν αρνούμαστε ε, για την υλοκτή Η αλυσίδα είναι μεγάλη, η αλυσίδα της υπεργολιβίας ορισμένες φορές είναι πολύ μεγάλη. Είναι υποχρεωτική ε, η κοινοποίηση των πληροφοριών πλέον βάσει της πρότασής μας για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το τονίζω όχι για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή προς το παρόν δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετά όριμη η κατάσταση για να έχουμε ένα πιο ενιαίο πλαίσιο. Ίσως στο μέλλον, ίσως σε μια δεύτερη φάση. Και αφού έχουμε κατοχυρώσει ότι και οι ίδιες επιχειρήσεις θεωρούν επωφελή την κοινοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Υπάρχουν και κατευθυντήρες γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις το Global Compact, την Παγκόσμια Συμφωνία του ΟΗΕ. Προβλέπονται δηλαδή σε άλλα διεθνή πλαίσια τέτοιες απαιτήσει. Έχουμε τον κώδικα βιωσιμότητας στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη. Ε, όμως εμείς δεν κρίνουμε ότι η έλλειψη πλαισίου θα δημιουργήσει πρόβλημα συγκρισιμότητας δεδομένων. Εξάλλου, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τις επιχειρησιακές πρακτικές τους ε, ε, θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις και με τις νέες πληροφορίες θα λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις ενισχύοντας έτσι de facto τη συγκρισιμότητα στην ενιαία αγορά. E Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδελφούς για τις ε, παρατηρήσεις. Θα ήθελα μόνο να επανέλθω σε δύο ζητήματα. Το γεγονός ότι ε, ε, δεν ενθουσιάζει αυτό το θέμα Ε, και δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι στο ευρωπαϊκό παραγωγικό σύστημα ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 500 εργαζόμενοι είναι μικρή επιχείρηση. Το θέμα δεν είναι μόνο ασυμμετρία ε, και ε, οι οικονομικές πληροφορίες και όλες αυτές που έρχονται να προσθεθούν Το θέμα είναι ότι όταν είναι εθελοντικό το σύστημα είναι κάτι το οποίο διαστρεβλώνει την εικόνα, αλλοιώνει το σύστημα και ακόμα και την ιδέα του τι είναι στη μικρομεσαία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη ε, ε, διάσταση, που είναι τόσο μεγάλες δηλαδή, ε, ε, έχουν ένα κρίσιμο μέγεθος που μπορούν να συλλέγουν και να διαβιβάζουν αυτά τα στοιχεία. Ούτε θα πρέπει να μας τρομάζει αυτή η υποχρέωση. Έχουμε και αρκετές προθεσμίες και διαδικασίες που είναι γνωστές τα τελευταία χρόνια. Και η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική πλέον και στους επενδυτές και στους καταναλωτές και θέλουν και οι δύο αυτές ομάδες να βλέπουν ποια είναι η ευθύνη της επιχείρησης, ε, πώς φέρεται μια επιχείρηση ως προς την κοινωνική της εταιρική ευθύνη, ως προς το περιβάλλον κτλ. Αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Στο παρελθόν δεν υπήρχαν τέτοιες απαιτήσει. Σήμερα οι καταναλωτές έχουν και αγοραστική αξία και μέσα στη διάθεσή τους και αγοραστική δύναμη δηλαδή και μπορούν να ελέγχουν τι κάνει κάθε εταιρεία και θέλουν πραγματικά να τα γνωρίζουν αυτά τα θέματα. Στο παρελθόν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον από πλευρά των καταναλωτών. Και το μόνο που ενδιέφερε τις επιχειρήσεις ε, ήταν η απόδοση των επενδύσεών τους. Ενώ τώρα ο κόσμος ενδιαφέρεται για περισσότερα πράγματα και ακόμα και οι ίδιες εταιρείες θέλουν να έχουν θετική εικόνα και υπεύθυνη εικόνα. Και οι ίδιοι επενδυτές επίσης δεν πρόκειται να επενδύουν σε μια επιχείρηση ε, που είναι πολύ επισφαλής εκτός αν θέλουν να βγάλουν πολλά λεφτά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι λοιπόν ε, μια θετική προσπάθεια αυτή η οδηγία και δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο φοβικοί. Είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος σίγουρα. Το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένως. Πρέπει να σας πω ότι έχω και επαγγελματική εμπειρία σε αυτό τον κλάδο εγώ. Θέλουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα σύστημα ενιαίο. Ε, μπορεί να υπάρχει πολλής δρόμος και ε, μεγάλες οι αντιστάσεις. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνειδητοποίηση των καταναλωτών για να επιλέγουν με τα λόγου γνώσεως. Αλλά να υπάρχει και μια θετική έτσι, ρύθμιση κάπως της αγοράς και μια προστιθέμενη αξία για τις ίδιες τις εταιρείε. Οι εταιρείε ανταγωνίζονται μεταξύ τους και καλό είναι να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη γνώση και πληροφόρηση. Είναι θετικό. Είναι άμυλα αυτό, δεν είναι ανταγωνισμός. Ε, υπάρχει το εξή παράδοξο. Οι εταιρείε που έχουν την καλύτερη συμπεριφορά γιατί σέβονται το περιβάλλον, γιατί σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ατομικά, έχουν και πλεονεκτήματα που αποκομίζουν από αυτή του την ενάρετη συμπεριφορά. Θα με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ να βρούμε κάποιες λύσεις συμβιβαστικέ. Ε, άρχισε η συζήτηση, δεν σταματά εδώ, θα συνεχιστεί και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αίσιο πέρας και να κάνουμε κάποια βήματα πρόοδου σε αυτό το δύσκολο δρόμο και μακρύ που μας περιμένει. Και όσο γίνεται να είμαστε πιο θετικοί αυτή τη στιγμή σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις ε, τροπολογίες σας, θα τις συζητήσουμε μαζί, κυρίως τις συμβαστικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν και κλείνει και αυτό το θέμα. Και 10 λεπτά νωρίτερα, ελπίζω αυτό να μην δυσκολεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα περάσουμε στην έκθεση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Παρουσίαση τη εκτίμηση επτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Παρευρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να περιμένουμε. Diamo 10 minuti. I tempi è anche indicato sono dati ogni mm. solamente puro, eh, pura indicazione, non è che sia Vi chiedo... Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα πέντε λεπτά υπομονή να κάνετε. Περιμένουμε να καταφθάσουν οι πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που είχαν ειδοποιηθεί για τις 5.30 για μας είναι ενδεικτικέ αυτές οι ώρες, αλλά εκείνοι τις θεωρούν δεσμευτικές και απόλυτες. Πριν τις 5.30 δεν έρχεται κανείς. Περιμένουμε 5 λεπτά και συνεχίζουμε στις 5.30. O arrivi, se uno solo, una sola, Λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο, δεν ξέρω και πόσοι θα έρθουν. Λίγα λεπτά υπομονή. Bene, Καλώς ορίσατε και πάλι μπορούμε να συνεχίσουμε διότι οι εκπρόσωποι της Επιτροπής ήρθαν. Σας καλωσορίζω. Χαιρετίζω και ακούμε τον Κάμιλ Κιλιάνσκι που θα σας παρουσιάσει την αξιολόγηση αντικτύπου για την οποία κάνουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Σα ευχαριστώ. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη από ό,τι φαίνεται είναι λάθος, Είναι λάθος από την πλευρά μας να θεωρήσουμε ακριβείς τι ώρες που αναφέρονται στην ημερησία διάταξη. 15 λεπτά φανταζόμαι θα χρειαστώ για την παρουσίαση. 10 διαφάνειες έχω ετοιμάσει και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω με ποιο σκεπτικό η Επιτροπή ε, προτείνει αυτή την, πρόταση και επίσης το περιεχόμενο της, την πρόταση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Ωραία. Ποια είναι τα κίνητρα της Επιτροπής. Γιατί το προτείνουμε. Κατά μία έννοια είναι προφανές. Οδηγεί σε σημαντική μείωση του κόστους και απλοποίηση των διαδικασιών ελαφρύνει το διαχειριστικό ε, άχθος όσον αφορά την τιμολόγηση. Αυτό προφανώς ε, θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διευκολύνει και ενισχύει την διαφάνεια και τη λογοδοσία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και επίσης εξίσου σημαντικά είναι και τα περιβαλλοντικά ωφέλη. όταν ανακοινώσαμε αυτή την πρωτοβουλία, πολύ ενδιαφερόμενοι εξεδήλωσαν το, το ενδιαφέρον τους και ε, αυτό εντάσσεται στην γενικότερη ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψηφιακό θεματολόγιο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αν και είναι κάπως προφανές ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα. Μας ανησυχεί η πιθανότητα κράτη-μέλη να προχωρήσουν χωρίς ε, συντονισμό και αυτό να δημιουργήσει πολλά και διαφορετικά πρότυπα που θα ανταγωνίζονται το ένα μεταξύ τους. Θα τα εξηγήσω λίγο περισσότερο αργότερα. Το πολιτικό πλαίσιο τώρα. Έχουμε την πολιτική υποστήριξη του Συμβουλίου η οποία εκφράστηκε τον Ιούνιο του 2012. το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 12, Επίσης ήταν ένα από ε, τα, σημεία κλειδιά της ε, πράξης για την εννέα αγορά 2 και συμπεριλαμβάνεται μια αναφορά σε αυτή την πρωτοβουλία και στην ετήσια ε, έκθεση ε, ανάπτυξης. Ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση. Δεν πρόκειται μόνο για μια διαβούλευση που έγινε μέσω ερωτηματολογίων. Οργανώσαμε επίσης και ε, ε, συγγνώμη, και συνέδρια για τις δημόσιες συμβάσεις γενικότερα και ειδικότερα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Γενικά υπάρχει έντονη υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας ε, ε της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πιστεύω ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα διαλειτουργικότητας είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση της δημόσιας συμβάσης. Έχουν ήδη αναλυφθεί διάφορες πρωτοβουλίες στο επιχειρησιακό επίπεδο, στο, επίπεδο της υλοποίησης. Έχουμε μια ανακοίνωση της Επιτροπής από το 2010. Υπάρχει ήδη ένα φόρουμ ε, πολυμερές των ενδιαφερομένων σε σχέση με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Υπάρχουν αναφορές σε αυτήν την πρωτοβουλία στην οδηγία για τον ΦΠΑ. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και διάφορα άλλα συγχρηματοδοτούματα, προγράμματα για την τιμολόγηση ε, ε, δημοσίων συμβάσεων. Γιατί αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία αυτή τώρα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι τόσο προφανές ότι είναι καλή ιδέα, αργά ή γρήγορα τα κράτη-μέλη θα αναλάμβαναν δράση, θα δημιουργούσαν σε εθνικό επίπεδο πλατφόρμες και προγράμματα δράσης, αλλά εάν συμβεί αυτό θα γίνει με τρόπο, ε, θα γίνει χωρίς συντονισμό. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα σύστημα που τελικά δεν θα είναι διαλειτουργικό. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας μεταξύ των διαφορών καθεστώτων και συστημάτων που εάν συνέβαινε αυτό θα είχαμε αρνητικό αντίκτυπο στις διασυνοριακές συναλλαγές. Εμείς θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν να δημιουργηθούν υπερβολικά πολύπλοκα συστήματα τα οποία δεν μπορούν να ε, ε, μιλούν το ένα μετάλλο, να είναι συμβατά το ένα μετάλλο αν, γιατί ένα τέτοιο, μια τέτοια κατάσταση θα δυσκόλευε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο της, του προσχεδίου οδηγίας. Το πεδίο εφαρμογή καλύπτει ε, την ηλεκτρονική τιμολόγηση μόνο όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και ε, οι δημόσιες συμβάσεις ορίζονται ε, στις τρεις σχετικές οδηγίες. Όμως καλύπτονται όλες οι ε, δημόσιες αρχές, αναθέτουσες αρχές σε όλα τα επίπεδα, το τοπικό, το περιφερειακό και το εθνικό. Θα αξιοποιήσουμε το CEN για να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις βελτιστές πρακτικές και στα ήδη υφιστάμενα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στα κράτη-μέλη. Ε, αυτό θα μας βοηθήσει επίσης να μην χρειαστεί ε, κράτη-μέλη που έχουν ήδη δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, που έχουν ήδη εφαρμόσει ηλεκτρονική τιμολόγηση, να αναγκαστούν να μεταβάλουν το σύστημά τους υπερβολικά. Θα ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ξεκινώντας από την άλλη άκρη, δηλαδή θα ε, διευκολύνουμε τους, τις αναθέτουσες αρχές να δέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Και προβλέπουμε μια μεταβατική περίοδο 4 ετών. Στην τελευταία διαφάνεια συνοψίζω μια, προ... μια πρόβλεψη για το μέλλον. Θεωρούμε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα υιοθετηθεί όλο και περισσότερο στο μέλλον. Αυτό φανταζόμαστε ότι θα αλλάξει και την συμπεριφορά των καταναλωτών και, θα, ε, και των ε, κρατικών αρχών και αυτό θα οδηγήσει σε ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γενικότερα. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην προσέλευση και ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις. Ε, παρακαλώ, η συνάδελφος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισκόπηση που μας δώσατε. Την περασμένη εβδομάδα ορίστηκα εισηγήτρια και μόλις την περασμένη εβδομάδα δηλαδή και είχα πολύ λίγο χρόνο να εμβαθύνω. Επί της αρχής μπορούμε να πούμε ότι είναι ευπρόσδεκτος ο στόχος και ε, ακριβώς ε, είναι σκόπιμο να εναρμονίσουμε κάπως την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και χαίρομαι που είναι σύντομο το κείμενο, 9 άρθρα μόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο ο δρόμος που προτείνεται είναι σωστός. Ο στόχος ναι, αλλά ίσως θα ήταν καλύτερο να θεσπιστούν κριτήρια για τις κοινοτικές προδιαγραφές για να γνωρίζουμε από εκεί και πέρα πώς μπορούν να εφαρμοστούν από τις διάφορες διοικήσεις και να κριθούμε από το αποτέλεσμα και να είναι το αποτέλεσμα ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει πλέον εκτήματα. Τώρα θα δείξει αν θα επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δέχομαι, αλλά θα προσπαθήσω κάποια πρότυπα να θέσω για να γνωρίσω γνωρίζουμε περίπου ποιο είναι ο γνώμονα και πώ θα μετρηθούμε και τι πρέπει να συντονίσουμε και να εναρμονίσουμε. Σε ορισμένες χώρε, όπως δείχνει η επισκόπησή σα, υπάρχει μια πρώτη διαδικασία Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία και Ιταλία είναι στα Σπάργανα. Για τη Γερμανία υπάρχει ε, με τις μεγάλες επιχειρήσεις έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια καλό θα ήταν να διδαχθούμε από την εμπειρία για να μην σε επιβαρύνουμε ιδιαίτερα. 48 μήνες είναι η προθεσμία για την εφαρμογή μου. Φαίνεται μικρό διάστημα αυτό, πολύ μικρό. Είναι υπερφιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα. Σε 14 μέρες λέει θέλετε να έχω την έκθεσή μου. Αυτή την εβδομάδα έχω δύο συνομιλίες για αυτό το θέμα. Την άλλη εβδομάδα είναι Στρασβούργο δεν ξέρω μπορώ να δεχθώ αυτή την προθεσμία 14 μέρες. Αν κάποιος θέλει να εργαστεί σοβαρά για ένα θέμα θα πρέπει να έχει και το χρόνο του να έχει τις απαραίτητες επαφές και συνομιλίες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Γνωρίζω ε, τις χρονικές υποχρεώσεις και τις συζητήσεις αλλά θα πρέπει να κάνουμε και σοβαρή δουλειά. Αλλά με κάθε σεβασμό τώρα 14 μέρες παρά είναι φιλόδοξο χρονοδιαγράμμα. Θα σας πω μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αν μπορώ να το δεχτώ ή όχι αυτό το χρονικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε, θέλω να πει κάτι. Θέλω να πω στην κυρία Κόλλιν Λάγκεν ε, ρητάω ότι θα την υποστηρίξω και χαίρομαι για τη συνεργασία που ήταν παγίως ε, πολύ καλή και θα κοιτάξουμε από κοινού πώς θα μπορέσουμε σε αυτό το στενό χρονικό κορσέ που μας έχουν βάλει ε, να το προλάβουμε. Ο Πρόεδρος. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση επ' ευκαιρία. Πολύ απλή και μπανάλα ίσως κοινότυπη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας υποθέσουμε, γιατί το έχετε ψάξει αυτό, ότι υπάρχει κάποια δυσκολία, καταλαβαίνω ότι υπάρχει, η χρήση αυτής της διαδικασίας μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις δεν μπορεί ενδεχομένω να φέρει μια μεγάλη αντίφαση Ξέρω ότι ε, ε, κινούμαστε από εταιρείε που έχουν πολύ μεγάλο πεδίο δραστηριοτήτων. Και επιβάλλουμε τώρα διαφορετική ε, διαδικασία στην άσκηση των εργασιών τους. Δεν θα ήταν ίσως καλύτερο να σκεφτούμε να εισαχθεί αυτή η διαδικασία για όλες τις συμβάσεις, είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές. Γιατί μόνο για τα δημόσια έργα. Δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι συνάδελφοι. Μήπω θα θέλατε να μα απαντήσετε στι ερωτήσει που σα έγινα. Ευχαριστώ πολύ εύλογα τα ερωτήματα. Ανέκαθεν υιοθετούσαμε τη σταδιακή προσέγγιση. Όντω αυτό επισύρει και κόστο κόστος μετάβασης. Κάποιες επιχειρήσεις ταυτόχρονα θα έχουν πολλαπλά συστήματα υποχρεωτικά. Αλλά δεν γίνεται ε, μία νυχτή να επιβάλλουμε τέτοιες ριζικές αλλαγές στην οικονομία και να ε, χρησιμοποιήσουμε τη σύνταξη σε δηλαδή να ενοποιήσουμε την πλατφόρμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε καν νομική βάση ούτως ή άλλως για τέτοιες προμήθειες, ε, γιατί ούτω ή άλλω επηρεάζεται ολόκληρη ή αλλω επηρεάζεται ολοκληρή πραγματική οικονομία και όχι μόνο οι κρατικέ προμήθειε. γιατί κάθε επιχείρηση έχει τα δικά τη πρότυπα και ούτω ή άλλω θα κάνει εξωτερική ανάθεση. Ε, πέρα από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ε, αληθεύει αυτό που είπατε ότι θα έχουμε κόστος μετάβασης καθώς και πολλαπλά αισθήματα που θα λειτουργούν ταυτόχρονα σε κάποιες επιχείρησεις για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν το αρνούμαστε. Προέδρο, πολύ ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω σε... Ε, στους παρόντες αλλά και σε όσους μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της εισηγήτριας. Τέσσερις και 5 Νοεμβρίου πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 7η Νοεμβρίου. 27 και 28 Νοεμβρίου θα συζητηθούν συμβαστικέ τροπολογίες. 16 Δεκεμβρίου θα συζητήσουμε για την συμβαστική πρόταση και στις 17 Δεκεμβρίου ε, προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ πιεστικό το χρονοδιάγραμμα. Συνήθω έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο. Βεβαίω, η συναδέλφοι θα αποφασίσει αν θα δεχτεί ή όχι το χρονοδιάγραμμα. Αυτά προβλέπονται πάντως για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ τους συναδέλφους που έμειναν εδώ μέχρι τελευταία στιγμή μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας 14 Οκτωβρίου το απόγευμα 3 με 6.30 θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Καλό βράδυ σε όλους. Σας